Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ. Κυρίσω την έναρξη της ε, συντακτικής συνεδρίασης, ε, τη συνεδρία συγκρότησης ΣΟΜΑ, της ε, Επιτροπής Μεταφορών. Θα προβούμε στην εκλογή του Προέδρου και τεσσάρων αντιπροέδρων. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στα αναπληρωματικά μέλη που μπορούν ε, να ψηφίσουν για το ΕΛΚ, ο κύριος Μαρινέσκου, ε, από τον κύριο Πρέντα, ο κύριος Μιζολέ από τον κύριο Προύστο, για την κυρία Λουκατσίγεβα δεν έχουμε ενημερωθεί. Για το ECR ο κύριος Βαντάλιν από τον κύριο Πραμπούν, ο κύριος Πορεμπά από τον κύριο Πιεσάχ και ο κύριος Πιοτρόφσκι από τον κύριο Κίρχαουπ. Για την ΚΟΕ, ο κύριος Φιναρέγιο από την κυρία Κόνεκα, ο κύριος Κατρούγκαλος από τον κύριο Ντεμεσί. Για τους σοσιαλιστές ο κύριος Ζέμκε από την κυρία Σενάλογα Έχουμε παληθεύσει την απαρτία, έχουμε υπερβεί κατά πολύ το 1 τέταρτο των μελών και παρακαλώ να υποβάλλετε τις υποψηφιότητες για την Προεδρία της Επιτροπής Μεταφορών. Κυρία Ντελή από πλευράς των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματος της ομάδας μου με χαρά ανακοινώνω την υποψηφιότητα του συναδέλφου Μίχαελ Κράμερ. Είναι ε, ένας ευρωβουλευτής που έχει καταδείξει πάθος και αφοσίωση για το έργο της Επιτροπής των Μεταφορών. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα όλοι σας να αναγνωρίσετε το έργο του. Δέκα χρόνια υπηρετεί εδώ στην Επιτροπή και επιθυμούμε να αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Σας ευχαριστώ. Δέχεται ο κύριος Κράμερ την υποψηφιότητα. Δέχομαι. Έχουμε επαληθεύσει ότι πληρούνται και προϋποθέσεις. Υπάρχουν άλλοι Υποψήφιοι για την Προεδρία. Όχι. Δυνάμει το κανονισμού, εάν δεν υπάρξει κάποια ένσταση, σας προτείνω διαβοής να εκλέξουμε τον Πρόεδρο. Σ' όλων, τον συγχαίρω, του εύχομαι μια επιτυχημένη και μακρά Προεδρία και τον καλό να έρθει να με αντικαταστήσει εδώ στο Προεδρείο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ασυνήθιστο τώρα για μένα να κάθομαι εδώ πάνω και να σας βλέπω κάτω εσάς από μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και ελπίζω να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία που είχαμε στην περασμένη θητεία και βεβαίως πάντα και με τη γραμματεία που υποστήριξε πάντα τη δουλειά μας. Ευχαριστώ και πάλι για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό μου και θα παρακαλούσα τις υποψηφιότητες σας τώρα για την πρώτη αντιπροεδρία. Από πλευρά των φιλελευθέρων, συγχαρητήρια Μιχαήλ Κράμερ για την εκλογή σα και εγώ προσβλέπω στην καλή συνεργασία και θέλω ω πρώτο αντιπρόεδρο να προτείνω τον κύριο Ντομινίκ Κρικέ ο οποίο είναι πάρα πολύ έμπειρο και στην Επιτροπή Μεταφορών και για όλου του παλιού βουλευτέ είναι πάρα πολύ ε, γνώριμο και γνωστό. Ελπίζω και να τον υπερψηφίσετε. Ναι, πολύ γνωστό είναι. Τώρα εδώ καθόταν ο κύριο Ζήκε. Λοιπόν, και το ξέρω και εγώ βέβαια ε, από παλιά. Υπάρχουν άλλε υποψηφιότητε. Όχι. Και εμεί διαβοή λοιπόν τότε να εκλέξουμε τον κύριο Ντομινίκ Ρικέ. Και να ξαναρωτήσω τον κύριο Ντομινίκ Ρικέ αν συμφωνεί. Ο οποίο έχει ήδη σηκωθεί βέβαια. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Και τον παρακαλώ να έρθει στο Προεδρείο και να λάβει τη θέση του. Ja, Δεύτερη θέση αντιπροέδρου. Παρακαλώ. Πρόταση έχουμε ο κύριος Βανακάμπ. Ναι κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να προτείνω το συνάδελφο Ντίτερ Λίμπρεχτ Κόχ, ο οποίος είναι και αυτός παλιά καραβάνα εδώ στην Επιτροπή. Εγώ είμαι νέο μέλος και μπορεί να με βοηθήσει πάρα πολύ. Προτείνουμε τον κύριο Κόχ λοιπόν ως δεύτερο αντιπρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φανακάμπ. Έχουμε υποψηφιότητα άλλη, εναλλακτική απέναντι. Παρακαλώ, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κόχ αν αποδέχεται αυτή την υποψηφιότητα. Ναι, με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Ωραία. Και πάλι διαβοής παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Κόχ, ελάτε να καθίσετε και εσείς στο Προεδρείο. Εσείς το ξέρετε λίγο καλύτερα από μένα το Προεδρείο. Και ερχόμαστε τώρα στον τρίτο αντιπρόεδρο. Παρακαλώ. Ναι. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Μικαέλ, τον Ντομινί και τον Ντίτερ για τις θέσεις ε, που αναλάβατε από πλευρά CCR. Ο Τόμας Πορέμπερ είναι ο υποψήφιος μας ε, για την Αντιπροεδρία. Δέχεται, είναι απόν αλλά μου διεμήνυσε να σας πω ότι δέχεται να ε, καταλάβει αυτό το αξίωμα. Αν το εκλεγεί. Μάλιστα. Έχουμε άλλη υποψηφιότητα εδώ. Όχι. Είναι δηλωμένη η συνένεσή του και η συμφωνία. Παρακαλώ διαβοής και πάλι να τον εκλέξουμε. Ο κύριος Τόμας Πορέμπα εκλέγεται λοιπόν και ερχόμαστε στον τέταρτο αντιπρόεδρο. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι υποψήφιος. Yes, thank you. Thank you, chairman. Uh, Ευχαριστώ. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την νέα σα θέση και συγχαρητήρια και στον αντιπρόεδρος. Ο υποψήφιο μας είναι ο Ούγγρος συνάδελφος Ιστβαν Ουιχιέλη. Δεν ε, καινούριος ευρωβουλευτής. Είναι εμπειρογνώμων σε θέματα τουρισμού και μεταφορών. Ήθελα να υποστηρίξετε την υποψηφιότητά του και να τον υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ. Άλλη υποψηφιότητα. Όχι. Όχι, εγώ είμαι ο Ιστβαν. Σηκώνω το χέρι μου για να με δείτε. με χαρά να συνεργαστώ μαζί σας στο Προεδρείο. Ωραία. Και πάλι διαβοής. Συμφωνούμε να τον εκλέξουμε. Das ist der Fall, dann bitte Μάλιστα. Παρακαλώ λοιπόν τον κύριο Ιστβαν να έρθει εκείνο στο Προεδρείο να καταλάβει τη θέση του. Okay, ja. Πολύ γρήγορα τα διεκπαιρεώσαμε και χωρί τριβή στην Επιτροπή μα Δεν θα είναι πάντα έτσι, έχουμε και διαφωνίε, αλλά εκεί είναι και το ενδιαφέρον και το συναρπαστικό πώς θα κάνουμε τη συζήτηση. Στην Επιτροπή Μεταφορών μας απασχολεί και οι μεταφορές και η κλιματική αλλαγή. Και μέχρι το 2020 επιβάλαμε ένα συνολικό ε, στόχο εκπομπών και για τις μεταφορές κατά 20% μείωση μέχρι το 2020 σε σχέση με τα στοιχεία του 90. Πολύ φιλόδοξο. Εδώ στην Επιτροπή μας πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία και γνωρίζουμε ότι αν δεν αλλάξει ο τρόπος ε, των συγκοινωνιών και των μεταφορών δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό γιατί από το 1990 κυρίως ε, στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 32% εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, στα νοικοκυριά 24% και στην ενέργεια 14%. Ταυτόχρονα στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές αυξήθηκε κατά 28%. Αυτό τι σημαίνει, αυτό ε, που πετύχαμε με δισεκατομμύρια χρήματα των πολιτών σε άλλους τομείς θα πρέπει να το επιβάλλουμε και στις μεταφορές διότι αυτό που κερδίσαμε απαλού χάθηκε διπλά και τριπλά στις μεταφορές. Καλή κινητικότητα ποιότητα βεβαίως να είναι δεδομένη να κυκλοφορεί ο κόσμος αλλά και το κλίμα να προστατεύεται. Επίσης δεν είναι επίμαχο ούτε στα κράτη-μέλη ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να εσωτερικευθεί το εξωτερικό κόστος. Θα το βρούμε και αυτό μπροστά μας και εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε και κάτι άλλο ιδιαίτερα επίκαιρο είναι το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο που έχουμε πάρα πολλά θέματα, το έχουμε ήδη αποφασίσει για τη συνέχεια θα δοθεί και αυτά θα τα δούμε όλα στη συνεδρία της 22 Ιουλίου όπου και πάλι θα ακούσουμε τον Επίτροπο, τον κύριο Σιμ Κάλλας και βεβαίως και την Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου. Ε, ε, θα ε, είναι παρόν ο υπουργό για τις προγραμματικές δηλώσεις και παρακαλώ να είστε κι εσείς όλοι παρόντες. Εδώ θα πρέπει λίγο να συντομεύσουμε γιατί συνεχίζεται αυτή η διαδικασία με άλλες επιτροπές που συγκροτούνται σήμερα σε σώμα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την τόσο πολυπληθή σας παρουσία και για την ψήφο σας. είμαι πεπισμένος και ελπίζω ότι θα σταθούμε όλοι στο ύψος της εμπιστοσύνης που μας δείξετε. Ευχαριστώ πολύ. Λήξη συνεδρίασης. Ναι,